So, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, ich hoffe, Sie hatten eine erfreuliche. Συνάδελφοι, ελπίζω να ήταν καλό το μεσημερινό διάλειμμα. Εγώ και έφαγα και διασκέδασα. Γιατί δούλεψα σε υπηρεσίες, εξωτερικές υπηρεσίες με τον ε, διευθυντή της ΕΝΤΖΑ, τον Βίλεμ Ντερόιτερ. Όχι, όχι, ήταν πολύ ευχάριστη η συνομιλία, γιατί είχαμε και πιο δυσάρεστες ε, περιστάσεις πριν από δύο χρόνια, θα θυμάστε βέβαια. Αλλά επειδή δεν ε, μπόρεσα να σας ε, ξεζουμίσω, όπως ο πρόεδρος ή αντιπρόεδρος. Έχω εδώ το κουμπάκι μου όμως, έχω και το σφυράκι μου και σας προειδοποιώ, όταν θα περάσει ο χρόνος ε, ομιλίας σας, τα πραγματικά θα πρέπει να ολοκληρώνετε. Όχι, εντάξει, δεν θα πειράξω εδώ πέρα το κουμπί του μικροφόνου, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει η δυνατότητα. Την... Στο τέλος της προηγούμενης συνεδρίασης, ο Σαλβαδόρ, Όχι, Σαλβαδόρ. Κάναμε την εισαγωγή, κάναμε την παρουσίαση του επόμενου τμηματο Και τώρα θα μιλήσουν οι ομιλητές που έχω στην, ε, στο κατάλογο ομιλητών. Πρώτος ο κύριος Γιώργεν, μετά ο κύριος Μπέγκε. Κάνεις άλλος? You the third one. Yeah. Um, Τρίτος είστε. Ποια, Μπέγκε, Φρανσουά. Ράιμα. Αχ, Quatsch. Entschuldigung. Γιώργος. <laughs> Ναι, με μπερδεύτηκα λίγο. Ναι, είναι δύσκολο μετά από ένα καλό μεσημερινό διάλειμμα να τα ξαναβρούμε πάλι. Και εγώ πέρασα πολύ καλά με τους εκπροσώπους των λόμπι της Γεωργίας. Αλλά αυτό είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Για τις εξωτερικές δράσεις, να πω το εξής. Συμφωνώ με αυτά που μας παρουσίασε ο Σάλβαδορ και το πώς εκτιμά την κατάσταση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ότι ο τομέας αυτός ε, έχει χρόνια υποχρηματοδότηση. Αυτό είναι σαφές. Να προσθέσω μερικά στοιχεία. Ειδικότερα θεωρώ ότι η πολιτική γειτονία, όπως αναφέρθηκε ε, και η Διεύρυνση, δεν αποτελούν μόνο μία προτεραιότητα, αλλά την κατεξοχήν προτεραιότητα για την εξωτερική δράση. Ιδιαίτερα σε μία κατάσταση όπως η σημερινή, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ε, έντονη στην διατύπωση σε ό,τι αφορά την πολιτική γειτονία και τη διεύρυνση για την επόμενη το συνομικό πλαίσιο. Θα αντιμετωπίσουμε ασφαλώ κάποια θέματα διεύρυνση. Ιδιαίτερα τώρα που αντιμετωπίσουμε τα θέματα τη Βορείου Και εδώ να υπογραμμίσω ένα πρόβλημα. Χτες έγινε η πρώτη συνάντηση με την πρώτη ομάδα ε, παρακολούθησης για την κατάσταση της Νοτιού Μεσογείου και το βασικό θέμα συζήτησης ήταν η χρηματοδότηση διάφορων μέσων. Και εδώ να κοιτάξουμε και το πρόβλημα που ανέφερε ο κ. Μπέκερ σήμερα το πρωί. Ο κίνδυνος ότι τα κράτη-μέλη, αν θέλουν να χρηματοδοτήσουν νέους τομείς, θα επιλέξουν ε, διακυβερνητικές μεθόδους και όχι κοινοτική μέθοδο. Και αυτό ασφαλώ αποτελεί πρόβλημα και για την εξωτερική δράση. Όταν χθε εξετάσαμε την κατάσταση χρηματοδότηση για την Βόρειο Αφρική, ασφαλώ έχουμε και την πολιτική για την γειτονία, αλλά έχουμε και συζήτηση για την ε, ανακούφιση του χρέου, για τα νέα προγράμματα γεωργία, για την Βόρεια Αφρική, το BRD, το EBRD, τι τράπεζε αυτέ, ε, για την ε, ενίσχυση του προπολογισμού, για μια νέα χρηματοδότηση για την νέα κοινωνία των πολιτών χρηματοδότηση των ε, ανθρωπιστικών αναγκών, τεράστιος αριθμός μέσων που δεν είναι συντονισμένα. Κάποια διακυβερνητικά, κάποια μέσω του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο στρατηγικοί στην προσέγγιση μας για τη χρηματοδότηση αυτή. Επίσης αναφέρθηκε η... Θεωρώ ότι θα πρέπει να αναφερθεί η αιρεσιμότητα, η ανάγκη για δημοκρατία. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο αυστηροί, να μιλάμε για αιρεσιμότητα σε ό,τι αφορά την ηθαγένεια. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο Ένα σχόλιο επιτρέψτε μου μόνο. Ο Σαλβαδόρ αναφέρει τον ε, πληθυσμό που γυράσκει για την ε, μετανάστευση κτλ. Να είμαστε λίγο πιο θετικοί, γιατί ο πληθυσμός που γυράσκει και η μετανάστευση δεν αποτελούν μόνο Απειλέ, δεν αποτελούν μόνο κάτι αρνητικό. Ναι, αποτελούν μεν μία πρόκληση, αλλά και μία δυνατότητα για θετικέ εξέλιξεις ενδεχομένω. Ο κύριο Μπέγκε, ευχαριστώ να συμφωνήσω κι εγώ μιλώντα για το θέμα της ηθαγένεια, της Ένωσης και για τα μικρά προγράμματα της κατηγορίας 3α, 3β ως τώρα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα με προτεραιότητα την νεολαία και τον πολιτισμό που είναι πάρα πολύ σημαντικά για την αντίληψη της Ευρώπης και ουσιαστικά χρηματοδοτούνται με σχετικά περιορισμένα μέσα και πετυχάνουν πολλά σε, πολιτική, σε ευρωπαϊκή δέσμευση και σε ό,τι αφορά τη θεώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα της μετανάστευσης και σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες για τη Frontex, το Ταμείο για του Πρόσφυγες κτλ. Βρισκόμαστε σε μια φάση αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά την εκτίμηση του πώς ε, η Ευρώπη μπορεί να ε, γίνει αλληλέγγυα, να φανεί αλληλέγγυα σε ό,τι αφορά τις νέες προκλήσεις και πώς ε, μπορούμε με τον δέντα τρόπο και από κοινού να αντιδράσουμε βάσει και όσων προδιαγράφουν ε, οι συνθήκε και η, χάρτη η... των βασικών δικαιωμάτων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα πρέπει να, προσθέσουμε... να προσέξουμε επίσης με ποια μορφή και σε ό,τι αφορά τα τρέχοντα μέσα, αλλά και σε ό,τι αφορά ενδεχόμενα μέσα που θα είναι καινούρια, που δεν προβλέπονται σε ό,τι αφορά την ευελιξία θα, ποια μέσα θα βρούμε λοιπόν προκειμένου να μην υπάρχουν κρίσεις ε, επί σειρά μηνών και πέρα από όλες τις διπλωματικές ε, διαφορές που δυστυχώ υπάρχουν στην Ευρώπη βρεθούμε και σε μία ε, διαμάχη για τον προϋπολογισμό και τελικά να μας πάρει έξι μήνες να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα, σε μία συμφωνία. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό στον τομέα αυτό. Κατά τα άλλα, συμφωνώ με την χρονική υποχρηματοδότηση της κατηγορίας 4. Ε, θα πρέπει να υπάρξουν πολιτικές λύσεις και αυτό τι σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός ε, σε ό,τι αφορά την γρήγορη κινητοποίηση και δυνατότητε αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Νομίζω ότι είναι καλό επίσης ε, πώς αναφέρει ο ε, εισηγητή στο θέμα της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Ε, ίσως θα πρέπει να εμβαθύνουμε λίγο και να παραθέσουμε πιο πολλά στοιχεία. Δεν είναι δυνατόν οι εθνικές διπλωματικές αρχές να συνεχίζουν να ορίζουν ως το νούμερο 28 της, την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες και σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή πολιτική θα πρέπει να επιμείνουμε προκειμένου ο πληθωρισμός ε, των μέσων να λάβει ένα τέλος. Φυσικά η ενσωματώση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης πέρα των ε, μέσων DCI ε, υπάρχουν και οι εθνικές δραστηριότητες και έχουμε το θέμα το, της αλλαγής του κλίματος σε διακυβερνητικό επίπεδο. Υπάρχουν και οι διεθνείς υποχρεώσεις και επίσης ε, εν ώψη των εξελίξεων στην Βόρεια Αφρική έχουμε και θέματα υπολογισμού και προτεραιοτήτων και πρέπει να πω ότι δεν είμαι απόλυτα ικανοποιημένος με αυτά που συζητάει η Αρμόδια Επιτροπή εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα πρέπει να φροντίσουμε να είμαστε πιο συνεπείς σε ό,τι αφορά την δαπάνη των... Ε, και κλείνει το μικρόφωνο του μιλητή. Η πρόεδρος υποθέτουμε. Ναι, Πρέπει. Ένα λεπτό. Διακόπη το μικρόφωνο διακόπηκε και η πρόεδρος το πήρε και τέλος πάντων τώρα ε, ελέγχει ότι λειτουργεί. Αλλά ο μιλητής ε, αναγκάστηκε να διακόψει. Φρανσουά. Ο Φρανσουά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Για το σημείο αυτό για την ηθαγένεια να ευχαριστήσω τον συγκεκριτή που σκέφτηκε να ευνοήσει την ε, ευρωπαϊκή επικοινότητα, την ευρωπαϊκή Επικοινόμορφια και τον ευχαριστώ. Σήμερα έχουμε ε, περίπου 20 γλώσσες και πολιτισμούς στην Ευρώπη που απειλούνται με εξαφάνιση. Και ε, υπάρχουν και κράτη όπως η Γαλλία, δυστυχώς που δεν δείχνουν το απαιτούμενο ενδιαφέρον. Πρέπει να επιμείνουμε από αυτού. Κάτι ακόμα. Μιλάτε για την ηθαγένεια. Καταρχήν στην Ευρώπη, μετά περνάμε στον υπόλοιπο κόσμο. Νομίζω ότι υπάρχει ένα κύκλος εδώ που θα πρέπει ε, ουσιαστικά να τον ε, χαρακτηρίσουμε. Υπάρχουν σημαντικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα. Σήμερα και στην οτιόχθη της Μεσογείου βρισκόμαστε ε, σε μια πρόκληση. είχαμε κάνει όσο έπρεπε πριν 20 χρόνια για τις χώρες της Ανατολής θα ήμασταν ε, σε διαφορετική κατάσταση σήμερα και με τη Λευκορωσία και ε, νομίζω ότι αν δεν αναλάβουμε δράση για όσοι συμβαίνουν σήμερα στην Ενότια οχθή της Μεσογείου θα μας ξεφύγει μια ιστορική ευκαιρία. Θα πρέπει να ε, επενδύσει η Ευρώπη σε μεγαλύτερη δημοκρατία και φυσικά αυτό θα μας οδηγήσει και σε λιγότερες μεταναστευτικές ροές. Ευχαριστώ. Ο Αλεξάνδρ. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ο εισηγητής ε, αναφέρθηκε στο θέμα της νομικής ασφάλειας, το οποίων άπτεται του ασύλου, της μετανάστευσης ε, και άλλων συναφών ε, θεμάτων. Ε, μέχρι το 2050 υπολογίζουμε ότι θα έχουμε 400 εκατομμύρια πρόσφυγες παγκοσμίως. 100 εκατομμύρια το χρόνο με, με υπολογισμούς Αυτά τα στοιχεία δεν νομίζω να επιβεβαιωθούν. Προέρχονται όμως αυτοί οι υπολογισμοί εδώ από το σώμα, άρα πολλοί έξοδες δεν θα πέφτουν, δεν νομίζω. Μήπως λοιπόν εν ώψη αυτών των προβλέψεων πρέπει να επισημάνουμε τα κεφάλαια αυτά του προϋπολογισμού με τα οποία μπορούμε να χειριστούμε αυτό το θέμα, παραδείγματος χάρη η εταιρική σχέση και το σημείο τρία των προτάσεων του εισηγητή, η Ευρώπη στον κόσμο. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς ε, μπορούμε να εντοπίσουμε τα κατάλληλα κεφάλαια, τα κατάλληλα σημεία στον προϋπολογισμό για να μπορούμε να καλύψουμε αυτά τα θέματα. Θα χρειαστούμε ε, περισσότερα, περισσότερες πιστώσεις, αυξημένες πιστώσεις για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας ή να καλύψουμε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στη διαχείριση του κυβερνοχώρου, στην ε, προστασία δεδομένων και ούτω καθεξής. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη ανάγκη, ε, ιδίως σε τεχνολογικά θέματα και ψηφιακές ε, λειτουργίες, να προβλέψουμε το μέλλον. Για να μην μακρηγορήσω, θα καταλήξω λέγοντας ότι επειδή και η Επίτροπος μας υποστήριξε πάρα πολύ, πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε δύο ταμεία, δύο ειδικά ταμεία. Ένα για την ασφάλεια, ένα για τη μετανάστευση και αυτά να καλυφθούν με την κατάλληλη χρηματοδότηση. Θέλω να πω ότι το σημείο 2, η θαγένεια, δεν με ικανοποιεί, δεν συμφωνώ με αυτό, διότι γιατί να μπλέξουμε τη νεολαία, πολιτιστικές εκδηλώσεις, επικοινωνία και ελευθερία με το θέμα αυτό της ηθαγένειας στον προϋπολογισμό. Θα ήθελα λοιπόν να εξετάσουμε εκ νέου αν είναι λογικό να διατηρήσουμε αυτή τη διάταξη και ιδίω τα σημεία 3α και 3β. Η πρόεδρος. Πολύ ωραία, ευχαριστώ και ο Σαλβαντόρ θα μας ε, μιλήσει για να ολοκληρώσουμε αυτό το τμήμα της συζήτησης πριν μπούμε στο, ε, στο επόμενο θέμα που είναι η δομή και η διάρκεια. Το είπα ήδη το πρωί, αλλά μπορείς να το ξαναπείς, Σαλβαντόρ. Ο Σαλβαντόρ θα ολοκληρώσει στο τέλος, θα μιλήσει στην αρχή του επόμενου γύρου βεβαίως και εν συνεχεία με τη σειρά των συντονιστών ή των εκπροσώπων των ομάδων. Ο Ράιμερ, Ράιμερ θα μιλήσει ε, θα, θα μιλήσεις στην αρχή στο τέλος του γύρου της συζήτησης. Το τέλος, εντάξει, ωραία. Απλώς για να ξέρω τη σειρά. Ξέρετε λοιπόν τη σειρά πώς θα μιλήσουμε. Ο Σαλβαντόρ τώρα. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. το θέμα που έδειξε ο κ. για τη μεταναστευτική πολιτική. Έχουμε δύο μέρη. Όλοι οι ομιλητές, ο Αλβέρο Λάιμαρ και ο Γιώναν, θέτουν το θέμα της μετανάστευσης. Εγώ δεν το βλέπω ως απειλή, αλλά και το βλέπω ως απειλή. Δηλαδή, μια μεταναστευτική διαδικασία ε, αν δεν ε, χρηματοδοτηθεί κατάλληλα, δηλαδή θα θέσει πρόβλημα και στους μετανάστες αλλά και στην ίδια τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι θέμα ασφαλείας για όλο τον κόσμο, δηλαδή μια καλύτερη μεταναστευτική πολιτική στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα θέσει εφαρμογή αν υπάρχει καλή χρηματοδότηση. Έτσι νομίζω ότι και η παρέμβαση της κυρίας Μάλστρομ ήταν πολύ ενδεικτική στο Στρασβούργο. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να αυξήσουμε τον όγκο των ε, πόρων, των κονδυλίων, γιατί θα ήταν και πολύ δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά πρέπει να γίνει ένας εξορθολογισμός των τεσσάρων ταμείων και αυτά να συγχωνευτούν σε δύο ταμεία. Τώρα αυτό το πώς θα γίνει θα το δούμε, αλλά θέλουμε να έχουμε ένα, μια καλύτερη διαχείριση των δαπανών, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε καταρχήν τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές ε, ροές και επίσης να μην έχουμε ε, και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο. Τώρα, η προβολή αυτής της κατηγορίας θα θυμάστε ότι ένα θέμα είναι η προβολή των διάφορων πολιτικών στο εσωτερικό μιας δομής και κάτι διαφορετικό είναι οι δημοθετικές προτάσεις που το συναντεύουν αυτό και που τελικά καθορίζουν την ε, ποσότητα των δαπανών, το μέγεθος των δαπανών. Εγώ θεωρούσα ότι ήταν ενδιαφέρουσα και ελκυστική η ιδέα να βάλουμε από κοινού ε, την ηθαγένεια και το χώρο ελευθερίας ασφάλειας και δικαιοσύνη στην ίδια κατηγορία. Ακριβώς ε, για το εξής. Ε, γιατί τα θέματα της ηθαγένειας και ασφάλειας δεν σχετίζονται ακριβώς, δεν εντάσσονται στη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020. Έτσι λοιπόν εγώ επέλεξα να το διατηρήσω σε μια άλλη κατηγορία αυτά. Όμως ε, θέλαμε κατά κάποιο τρόπο να το συνδέσουμε αυτά τα θέματα με θέματα εσωτερικής δικαιοσύνης και την πολιτική γειτονία, γιατί σχετίζονται με τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Όμως το θεμελιώδες πρόβλημα όπου μπορεί να υπάρχει ένα σύνδεσμος μεταξύ πολιτική γειτονία και μεταναστευτική πολιτικής ε, είναι στη Βόρεια Αφρική. Δεν συμβαίνει το ίδιο με άλλες ε, περιοχές ε, που θίγονται από την πολιτική γειτονία. Έτσι λοιπόν, εγώ επί της αρχής, εκτός αν εσείς έχετε διαφορετική άποψη, θα προτιμούσα να αφήσω την ε, πολιτική γειτονία στην κατηγορία η Ευρώπη στον κόσμο και την κοινή μεταναστευτική πολιτική να παραμείνει στο χώρο ελευθερίας ασφαλής δικαιοσύνη και ηθαγένειας. Τώρα, αν ε, δεν χρειάζεται να υπάρξει αύξηση των κονδύλιων για την πολιτική γειτονία, αυτό θα ήθελα να το κρίνουν οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Ανάπτυξης και από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εγώ είμαι απλώς μέλος της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμών. Δεν ε, μπορώ να τοποθετηθώ για το πώς καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πολιτική γειτονίας. Όμως θεωρώ όπως και να έχει ότι η Βόρεια Αφρική είναι προτεραιότητα σημαντική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει και κάποιος δημοσιονομικός αντίκτυπος για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση στη Βόρεια Αφρική. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση, κατάλληλη χρηματοδότηση στην κατηγορία των εξωτερικών δράσεων. Το ίδιο ισχύει και για το αποθεματικό έκτακτης ανάγκης αφού συνάντησα την Επίτροπο, ε, την Αρμόδια Επίτροπο για την ε, Ανθρωπιστική Βοήθεια, τέθηκε αυτό το θέμα. Δεν ε, μπορεί τώρα το παθηματικό να ενεργοποιηθεί αμέσως, χρειάζεται συμφωνία του Συμβουλίου, χρειάζονται διαπραγματεύσεις και πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε γιατί αυτές οι ανθρωπιστικές κρίσεις ξεσπούν και πρέπει να αντιδράσουμε πολύ γρήγορα. Αν ε, έχουμε λοιπόν ε, τέτοιε περιπτώσει όπω έχουμε σήμερα στη Βορεια Αφρική, τέτοιου είδου κρίσει, τελικά τελειώνει ο προπολογισμό, τα κονδύλια που έχουν προβληθεί μέσα σε τρει μήνε και πρέπει να προσφύγουμε σε αυτό το αποθεματικό έκτακτη ανάγκη. Αυτέ τι δυσκολίε ε, αντιμετωπίσαμε στην κατηγορία των εξωτερικών δράσεων και γι' αυτό θα συμπεριλαμβάνω όλα αυτά στο αντίστοιχο κεφάλαιο. Αυτές είναι οι ανησυχίες που έχουμε, Πρόεδρε και βλέπω ότι συμπίπτουν με τις ανησυχίες που εξέφερσαν ορισμένοι εκ των συναδέλφων. vielen Dank. Ε, Ευχαριστώ. Εντάξει, δεν έχουμε μακρύ δρόμο να διανύσουμε, ε, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε με τον τρίτο γύρο, δηλαδή τη συζήτηση του τρίτου τμήματος, χρονική διάρκεια και ε, δομή, διάθρωση. διάρθρωση. Συγχωρείτε, είχα στα χαρτιά μου, λέει ο μιλητής. Τα βρήκα όμως τώρα. Λοιπόν, το τέταρτο τμήμα αναφέρεται γενικά σε τεχνικά ζητήματα. Ξεκινά από την παράγραφο 90 και φτάνει μέχρι το τέλος της έκθεσης. Μέχρι το σημείο 121. Εδώ περιλαμβάνονται πολλά τεχνικά ζητήματα αλλά και το ακαθόδε και λεπτό θέμα της μελλοντική χρηματοδότηση του μέγεθου του προπολογισμού και των ε, πιθανών μελλοντικών ιδιών πόρων. Ας ξεκινήσουμε με τη δομή. Η, πρότασή μου για τη δομή βασίζεται σε μια σειρά συμπερασμάτων που προσπάθησα να εξαγάγω από τις συζητήσεις που είχαμε στην Επιτροπή Σούρου όλους αυτούς τους μήνες. Ξέρω ότι είναι πολεμική, ότι είναι επίμαχη όπως ε, ε οποιαδήποτε άλλες από τις δομές που θα μπορούσε να παρουσιαστεί εδώ για το κείμενο. Έχω παρουσιάσει πολλές και το ξέρουν οι συνεργάτες μου. Έχουμε παρουσιάσει πάρα πολλές εναλλακτικέ ε, σε σχέση με τη δομή και είμαστε πολύ ευέλικτοι στην τροποποίηση της δομής του κειμένου. Γιατί τελικά μετά από κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής μας τροποποιήσαμε εκ νέου τη δομή γιατί θεωρούσαμε ότι μετακινούνταν η πλειοψηφία. Κάποια στιγμή φυσικά μπορεί να παρουσιάσω κάτι και να πω ορίστε αυτό παρουσιάζω τώρα και να δεχτώ και την ανάλογη κριτική. Όμως το θέμα είναι ότι θέλουμε να δώσουμε την απαραίτητη προβολή στη στρατηγική Ευρώπη 2020. Όλοι συμφωνούμε από αυτό νομίζω. Νομίζω ότι πρέπει να αποφύγουμε μια αυστηρή κατηγοριοποίηση των διάφορων πολιτικών ε, υπό τον ε, τίτλο της εφιούς ε, ή φόρου ανάπτυξης ή της καθολικής ανάπτυξης. Ε, πάντως είναι πολύ δύσκολο να εξεύρουμε ε, κάτι που να αφορά το περιεχόμενο του προϋπολογισμού ή ε, υπό τον τίτλο «Καθολική ανάπτυξη, συμπεριληπτική ανάπτυξη». Αν βρείτε εσείς κάτι, ευχαρίστως να μου το πείτε. Από την άλλη... Σα το είχα πει και στο παρελθόν. Όπω ε, λέει και ο συνάδελφο Ζεχαρτ Βάρμε, ίσω να είναι συντηρητική η δομή αυτή των δημοσιονομικών προοπτικών, όμως δεν θέλουμε να κάνουμε εδώ ριζικές αλλαγές. Γιατί δεν είμαστε και πολύ σίγουροι ότι θα υπήρχε επαρκής πλειοψηφία για να υποστηρίξει τέτοιες ριζικές αλλαγές. Αυτή η δομή πάνω κάτω λειτουργεί καλά πέρα των κριτικών. Εντάξει, υπάρχουν και μειονεκτήματα, προσπαθήσαμε να τα επιλύσουμε. Εγώ προτείνω λοιπόν μία δομή όπου ομαδοποιούμε όλους τους τομείς που συμπεριλαμβάνονται στη στρατηγική για το 2020 ως εσωτερικές πολιτικές με τρει υποκατηγορίες. Η πρώτη αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση, η δεύτερη την αηφόρο ανάπτυξη και η τρίτη την πολιτική συνοχής. Έχουμε εισαγάγει μια ξεχωριστή κατηγορία για την ηθαγένεια. Εδώ περιλαμβάνονται και τα θέματα εσωτερικής ασφάλειας. Τρίτη κατηγορία για τις εξωτερικές δράσεις για να εθετήσουμε και την αερολογία της αναθεώρησης. Λέμε Global Europe, η Ευρώπη στον κόσμο εδώ. Μια κατηγορία για την ε, διοίκηση. Και ως καινοτομία θέλουμε να παρουσιάσουμε τη χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση για να υπάρξει ένας πιθανός σύνδεσμος μεταξύ του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού με το μηχανισμό σταθερότητας μετά το 2013. Αυτό σχετίζεται στενά με κάτι για το οποίο δεν ξέρω αν υπάρχει συνένεση στην Επιτροπή να διατηρήσουμε την κοινοτική μέθοδο έναντι της διακυβερνητικής μεθόδου που νομίζω ότι δεν είναι καλή ούτε για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σύνολό τη και πολύ λιγότερο για τα συμφέροντα και τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή η νέα κατηγορία ε, υπόκειται σε οποιαδήποτε κριτική, όμως πιστεύω ότι ως πολιτική δήλωση για το τι επιθυμεί το Κοινοβούλιο είναι απαραίτητο να την αναγράφουμε. Διάρκεια. Αφού το αναλύσαμε, εις βάθος σκεφτήκαμε ότι το καλύτερο είναι να συνεχίσουμε με τα 7 έτη, τουλάχιστον για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο, γιατί δεν έχουμε καμία εγγυήση για το, η συμφωνία στην οποία θα καταλήξουν τα κράτη-μέλη. Θεωρούμε λοιπόν ότι τα 7 έτη μας επιτρέπουν ε, τουλάχιστον να διατηρήσουμε τα θετικά που είχαμε μέχρι τώρα μία επαρκή περίοδο προγραμματισμού για τις πολιτικές συνοχής, για την αγροτική πολιτική, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Δεν μας αρέσει το 5 συν 5 έτη ε, γιατί δεν ξέρουμε αν θα μπορούσε να υπάρξει μία μεσοπρόθεσμη ρήτρα αναθεώρηση. Έχουμε τέτοια εμπειρία από το Συμβούλιο και έτσι θεωρούμε ότι τα 7 έτη στις σημερινές συνθήκες είναι η καλύτερη δυνατή πρόταση. Και δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα στην ευελιξία. Γιατί έχουμε την εμπειρία για το πώς ε, λειτουργήσε η ευελιξία σε αυτές τις δημοσιονομικές προοπτικέ. Χωρίς περισσότερη ευελιξία στο σύστημα δεν μπορούμε να έχουμε μία ορθή εκτέλεση των επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών. Η σημερινή ευελιξία είναι ιδιαίτερα ελληπή. εξού και μεγάλο τμήμα των ε, συζητήσεων ε, θεσμικού χαρακτήρα που λαμβάνουν χώρα στην Επιτροπή Περιπολογισμών έχουν να κάνουν ε, με το διαφορετικό τρόπο που κατανοούν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο την έννοια της ευελιξίας. Εγώ στην έκθεση σας υποβάλλω ορισμένε προτάσεις. Καταρχήν, μια νομική δεσμευτική υποχρέωση για να υπάρξει μια μεσοπρόθεσμη ενδιάμεση αναθεώρηση, αναθεώρηση των ανώτατων ορίων και δεύτερον ενίσχυση της ευελιξίας ε, κάθε ενός από τα ανώτατα όρια με διάφορους τρόπους είτε με ένα τρόπο αναδίπλωσης είτε με ε, αύξηση της δυνατότητας μεταφορών μεταξύ των διάφορων κατηγοριών δαπανών είτε της μεταφοράς ε, των περιθωρίων που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από το ένα το στο άλλο, κάτι που νομικά είναι δυνατόν. Από την άλλη αναφέρουμε μια πλουστευμένη διαδικασία για την αναθεώρηση των πλαφών ε, κάτω από ένα συγκεκριμένο κατόφυλλο έχουμε το 0,03. Ξέρετε ότι αυτό είναι ένα προβληματικό σημείο με τις ε, διαπραγματεύσεις, με το Συμβουλίο και το Κοινοβούλιο. Θα θέλαμε βέβαια ένα μεγαλύτερο ποσοστό για αυτή την ευελιξία για το μέλλον. Και κατόπιν πιστεύουμε ότι πρέπει να ενισχυθεί το σημερινό σύστημα μηχανισμού ευελιξίας και για το μέσο για την ευελιξία, για τον χανισμό ευελιξίας, αλλά και για το αποθεματικό έκτο της ανάγκης, ε, όπως και για το Ταμείο Ολληλεγγύης και το Ταμείο Αντιμετώπισης της Παγκοσμιοποίησης. Πρέπει να βελτιώσουμε την εφαρμογή. Και επίσης ε, εκεί όπου έχουμε κάποια αποθεματικά που δεν έχουν ε, κατανεμηθεί ε, στα περιθώρια πρέπει να αντιμετωπιστεί και αυτό και επίσης πρέπει να δημιουργήσουμε πιθανά ε, μία και κονδύλια που θα ενεργοποιούνται πάντοτε μέσω της κοινοτική μεθόδους και θα ενεργοποιούνται μόνο όταν ε, κάποιες προϋποθέσεις που δεν έχουν προβλεφθεί εκ των προτέρων εμφανίζονται στον δημοσιονομικό προγραμματισμό. Την περισπασμένη θητεία είδαμε πριν το σχάρι το θέμα για ένα ταμείο για την ενέργεια. Δεν υπήρξε συμφωνία. Όμως ε, βλέπουμε ότι αυτά τα ad hoc ε, ταμεία ή κονδύλια για να αντιμετωπίσουν ορισμένες ανάγκες της Ένωσης ε, θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα. Χωρίς φυσικά να υπάρχει επίπτωση στις αιτήσιες δεσμεύσεις των κρατών μελών. Έχω μια αμφιβολία. Θέλετε να σταματήσω εδώ και κατόπιν να αναφερθούμε στο μέγεθο του προπολογισμού και στου ίδιου πόρου. Ναι, λέει η Πρόεδρος. Θα ασχοληθούμε με το ύψος του προϋπολογισμού ξανά στις 7 Απριλίου. Καλώς μέχρι εδώ και αυτά τα οποία είπες μέχρι τώρα για την προτινόμενη διάρθρωση είναι σωστή και είναι σημαντικό να έχουμε τέτοιες ε, άμεσες ε, εικόνες, ένα είδος Φωτογράφηση δηλαδή από το πριν και το μετά. Πώς ήταν η εικόνα παλιά, πώς ήμασταν <laughs> νεότεροι και πώς είμαστε τώρα. Μπορεί μάλιστα να διαπιστώσουμε ότι από τη μία φωτογραφία στην άλλη υπάρχει βελτίωση. Τα πράγματα έγιναν καλύτερα. Και δεν απορρίπτω κάπως μια πιο συντηρητική προσέγγιση, όπως το προείπε ο Ράιμερ, όταν λέω συντηρητικά, εννοώ με σταθερότητα αλλά και διάθεση για αλλαγή. Εγώ ως σοσιαλδημοκρατική βουλευτής από τη Βόρεια Ορεινανία Βεσφαλία δεν μπορώ να αρνηθώ μια πιο συντηρητική προσέγγιση. Εμείς ε, λέμε στη δική μου περιφέρεια ότι θέλουμε να προχωρήσουμε. Η σοσιαλδημοκρατία σημαίνει πρόοδος ε, με προσεκτικά βήματα. Η Έιντα. Uh, Eh, Ευχαριστώ. Νομίζω ότι έχω πέντε λεπτά. Θα προσπαθήσω να μπω στην ουσία. Όπως είπατε και εσείς, Πρόεδρε, η αναγκαιότητα να έχουμε μία δομή, μία διάρθρωση προέρχεται ακριβώ γιατί έχουμε μία φωτογραφία στιγμή που μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τη λογική των δαπανών ε, και να δούμε ποιες είναι οι πολιτικές προτεραιότητες, να αναδείξουμε τις πολιτικές προτεραιότητες που έχει το Κοινοβούλιο μαζί με το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Και το να έχουμε μια καλή δομή ικανή να κατοπτρίζει αυτές τις προτεραιότητες και να έχουμε αυτή τη φωτογραφία είναι σημαντικό. Και μέσα σε αυτή τη δομή είναι σημαντικό να έχουμε και κατηγορίες. Γιατί έχουμε αυτές τις κατηγορίες. Πιστεύω ότι η λειτουργία ε, είναι δυτή. Αφενός, γιατί το να έχουμε μια κατηγορία προστατεύονται αυτές οι δαπάνες, δηλαδή είναι προορισμένες προς ένα πολιτικό στόχο, αλλά ταυτόχρονα τίθεται και ένα πλαφόν, ένα ανώτατο όριο για τις δαπάνες. Και εκεί πρέπει να συνδυάσουμε μεταξύ της προστασίας μιας πολιτικής προτεραιότητας και συνεπώς μιας δαπάνης και του περιορισμού, του ορίου που θέτουμε σε αυτή την πολιτική. Έτσι λοιπόν, δεν ε, θα μπορούσαμε ε, να έχουμε εδώ μία δομή με δύο κατηγορίες ε, γιατί διαφορετικά θα, θα υπήρχε σαφήνεια στις ιδέες μας αλλά ούτε θα μπορούσαμε να δεκτούμε και μία πρόταση με 20 κατηγορίες γιατί δεν θα είχε και νόημα και κάτι ακόμη. Η δομή είναι σημαντική. Είναι σημαντική αυτή η σταθερή εικόνα, η σταθερή φωτογραφία, αλλά ε, κοιτάξτε, η δομή δεν θα σημάνει ότι αναλόγως με το είναι καλύτερη χειρότερη, θα είναι και καλύτερη χειρότερη και ε, η υλοποίηση, η εκτέλεση του προπολογισμού. Εμεί ε, γενικά μπορούμε να συμφωνήσουμε με την πρόταση του εισηγητή, αλλά με κάποιε αποχρώσεις. Το λέω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ένα μεγάλο βαθμό, γιατί πιστεύουμε ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 είναι κύρια προτεραιότητα και καλύπτει και μια σειρά πολιτικών όμω με αποχρώσει αποχρώσεις γιατί. Γιατί θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε αιμονή με αυτή την στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 σε σημείο που να υπάρχουν κάποιες ε, συνέπειες και να προσπαθήσουμε ε, κάποιες πολιτικές που δεν έχουν να κάνουν με τη στρατηγική για το 2020 να το βάλουμε κάτω από αυτή την ομπρέλα έτσι ώστε να φαίνεται ότι όλα ανήκουν εκεί. Θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε με κάποιες μικρές αποχρώσεις Αν και γενικά σας είπα, θα μπορούσαμε να την ε, δεκτούμε σε μεγάλο βαθμό αυτή τη δομή. έχουμε κάποια αμφιβολία σε σχέση με αυτή τη νέα κατηγορία χρηματοπιστωτικής διακυβέρνησης. Και από ό,τι καταλαβαίνω ότι υπάρχει σύνδεση εδώ με το μηχανισμό χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Φυσικά υπερασπίζουμε την κοινότητα και μέθοδο, αλλά δεν κατανοούμε πολύ καλά. Εδώ σε τι αναφέρεστε, μιλάτε για μια γραμμή προπολογισμού που, όπου θα είχαμε μια εγγύηση, δηλαδή μια γραμμή χωρίς χρήματα. Τελικά ποια είναι ακριβώς η ιδέα σας εδώ σε σχέση με την ευελιξία. Συμφωνούμε απόλυτα με τα θέματα αυτά. Φυσικά το θέμα της ε, ευελιξίας το συζητούμε εδώ και πολύ καιρό, όχι μόνο σε αυτή την Επιτροπή, αλλά και στην Επιτροπή Περιπολογισμών. Είναι ζωτική σημασία στο ζήτημα, αλλά είναι πολιτικής βούλησης επίσης. Μπορούμε να έχουμε ή ένα μέσο ευελιξίας ή χίλια, αλλά τελικά αν υπάρχει συμφωνία και αν υπάρχει πολιτική βούληση για την εφαρμογή, τότε θα το δούμε, δεν μπορούμε να έχουμε λιγότερες ή μικρότερες ε, δυνατότητες ευελιξίας. Το θέμα αυτό εξαρτάται από τη Βουλή, κυρίως του Συμβουλίου, να εφαρμόσει αυτό το μέσο. Σε σχέση με την ενδιάμεση αναθεώρηση. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα να προσπαθήσουμε να πετύχουμε αυτές τις ενδιάμεσες αναθεωρήσεις. Υποθέτω ότι μιλάμε για περιόδους 7 ή 10 ετών. Τα 5 έτη δεν νομίζω ότι θα ήταν μια λογική επιλογή. Για το θέμα της ευελιξίας συμφωνούμε και για τα περιθώρια τώρα. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Αλλά προσοχή, πώς υπολογίζονται τα περιθώρια αυτά, γιατί από τη δική μας άποψη, από τη δική μας σκοπιά, θα πρέπει να ξέρουμε τι δαπάνε ε, ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία και εκεί να προσθέσουμε το περιθώριο, όχι να ψάξουμε να ζητήσουμε τι συνολικέ δαπάνε και μετά να αφαιρέσουμε το περιθώριο να δούμε τι θα προσθέσουμε. Τώρα για τη διάρκεια εδώ έχουμε μια διαφοροποίηση γιατί για μας η διάρκεια του δημοσιονομικού πλαισίου είναι ένα δίλημα. Ή πρέπει να ξεβρούμε την ισορροπία μεταξύ τη σταθερότητα και τη προβλεψιμότητα ή των κοινοβουλευτικών θητιών. Και κατόπιν θα έρθει η ευελιξία. Όσο μεγαλύτερη διάρκεια, με τόσο μεγαλύτερη ευελιξία. Και γι' αυτό ή θα είναι ή 7 ε, ή 5 συν 5. Αν είναι 5 συν 5 θα πρέπει να δούμε πώς ε, θα το διαρθρώσουμε σε δύο εντολές ή αν θα γίνει κάποια επιμήκυνση. Jetzt kommt an Jensen. Ευχαριστώ. Αν Γιέντζεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ είχα προτείνει να μην έχουμε κατηγορίες. Καλό είναι να έχουμε μία ε, σαφή δομή στον προϋπολογισμό και καλό είναι επίσης, δέχομαι ε, να έχουμε μια σταθερότητα κάπως συντηρητική, αλλά μέσα στις κατηγορίες που υπήρχαν το είχαμε αυτό. Στην ένα αλφα παραδείγματος χάρη, οι πιστώσεις μεταφέρονταν από την έρευνα στις μεταφορές και ούτω κάθε εξής. Είναι ευκολότερο εάν ένα πρόγραμμα δεν είναι αποτελεσματικό να πάρουμε τα κονδύλια από αυτό και να τα δαπανίσουμε αλλού. Η μεταφορά ε, πιστώσεων μεταξύ κεφαλαίων είναι καλύτερα. Ε, ε, είναι, πιστεύω, ένα σωστό μέσο. Όσο όμως λιγότερα είναι τα κεφάλαια αυτά από τα οποία μεταφέρουμε, τόσο καλύτερα. Ούκεν το πολλό το εφ. Αυτές, αυτή τίτλοι που έχει τώρα ο Σαλβαντό στον πίνακά του ας πούμε είναι δυνατόν ε, να μεταφέρουμε πιστώσεις από τον ένα τίτλο στον άλλον 80% το βάζεις σε έναν τίτλο και εν συνεχεία διάφορους άλλους μικρότερους ε, Freedom, Security and Justice very much would like to Και δεν ξέρω αν σε αυτή τη διάταξη που έχεις είναι δυνατό να γίνουν αυτές οι μεταφορές. Ε, πρέπει να εξασφαλίσουμε την ευελιξία που χρειάζεται στην ε, διάθρωση αυτή για να εξασφαλίσουμε ε, την έκφραση του κυρίου Σέρτσεν για αλληλεγγύη και ασφάλεια και σταθερότητα βεβαίως. Αυτά τα στοιχεία χρειάζονται στην αντιμετώπιση της μετανάστευσης, της ε, συνεργασίας, ε, στο άσυλο κλπ. Είναι στοιχεία της πολιτικής καλής γυτνίασης. Εν κατακλείδη αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να έχουμε λιγότερα, ε, λιγότερα κεφάλαια στον προϋπολογισμό ή λιγότερους το μίσο στον προϋπολογισμό, διότι έτσι θα μπορέσουν πιο εύκολα οι αρμόδιοι επί της γεωργίας να υπολογίσουν ποια χρήματα, ποια ποιες πιστώσεις θα επιστραφούν για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν αλλού. Το πρόβλημα όμως δεν είναι η επιστροφή των χρημάτων για επαναχρησιμοποίηση. Το πρόβλημα, το, ο στόχος ο δικός μας είναι ευελιξία στη διαχείριση των πιστώσεων. Όσον αφορά την διάρκεια των δημοσιονομικών προοπτικών, προοπτικών, η ομάδα μου προτιμάει τα πέντε χρόνια. Μπορούμε να δεχτούμε όμως 7 ως μεταβατικό στάδιο, διότι ε, αν την επόμενη φορά εφαρμόσουμε την πενταετία, θα βρεθούμε σε μία ε, ανόητη κατάσταση, με μία νέα ε, νεοεκλεγή σε επιτροπή, ένα νεοεκλεγέν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν θα είναι δυνατόν να λειτουργήσει έτσι. Καλό είναι λοιπόν να αποφασίσουμε την εφταετή περίοδο. Μετά όμως να προσθέσουμε ότι μετά από τα 7 αυτά χρόνια θα συνεχίσουμε με πενταετής περιόδους, ίσως 5 συν 5 για τα διαφορετικά ταμεία ή μακροπρόθεσμα προγράμματα. Η γενική αρχή θα πρέπει να είναι κάθε νομοθέτης του Κοινοβουλίου και κάθε εκτελεστική επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τις δημοσιονομικές προοπτικές. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μετακινηθούμε στο μέλλον σε πενταετές περιόδους. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπερασπίσουμε και να κοιτάξουμε να επιβληθεί. Να το επιβάλλουμε με κάθε προσπάθεια εκτός από την επόμενη περίοδο που πιστεύω μπορεί να είναι 7 Θα κάνουμε τις αντίστοιχες διαβουλεύσεις βέβαια και με το Συμβούλιο. Επίσης, ε, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέει ο, Σαλβατόρ με τα μέσα ευελιξίας. Ε, Πρέπει να σκεφτούμε αν χρειαζόμαστε νέα ή αν πρέπει τα υπάρχοντα να προσαρμοστούν. Οπωσδήποτε πρέπει να έχουμε ευελιξία. Και εάν υιοθετήσουμε κατηγορίες και περισσότερες κατηγορίες, τόσο πιο πολύ ευελιξία θα χρειαστούμε. Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ Σαλβαντόρ. Και ε, έτσι μπορούμε να έχουμε ένα θαυμάσιο έναυσμα και για τις δικές μας συζητήσεις. Ε, είναι ένα κάλεσμα που μας οδηγεί προς την κατεύθυνση την οποία έχουμε και εμείς κατά νου. Καταρχάς για τη διάρθρωση είναι ενδιαφέρον, αν κοιτάξουμε αυτό τον ε, πρώτο, το πρώτο τίτλο, 85 με 95% α, είναι στο πρώτο, στο πρώτο κεφάλαιο, στο πρώτο κεφάλαιο, το οποίο έχει τίτλο ε, «Ανάπτυξη, ε, ε, ολοκληρωμένη ανάπτυξη». Και αυτό ο πρώτος, το, το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει το 90% του προϋπολογισμού. Αυτοί οι στόχοι τους οποίους θέτουμε για το 2020 είναι ευρύς. Ε, για την εφορία, την ε, ολοκλήρωση, τη συμπερίληψη, τον μη αποκλεισμό, την ε, συνετή διαχείριση κλπ. Τουλάχιστον στο πρώτο κεφάλαιο η αηφόρος ανάπτυξη καλύπτεται και εν συνεχεία στους διάφορους τίτλους έχουμε την, το γεωργικό κεφάλαιο, το αλληλευτικό κεφάλαιο και λοιπά. Αυτό που πρέπει πιστεύουμε να διαχωρίσουμε σε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο είναι ε, η έρευνα και ανάπτυξη. Έχουμε πει επανειλημμένως ότι η Ευρώπη πρέπει να προωθήσει την έρευνα και την ανάπτυξη. Άρα λοιπόν χρειάζεται το R&D, ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, καινοτομική έρευνα, ανάπτυξη και ούτω καθεξής. Τώρα, συνοχή, συνοχή, ε, η περιφερειακή συνοχή, ε, το θέμα της ηθαγένειας και αυτό είναι πολύ ωραία, άλλο κεφάλαιο. Εν συνεχεία το τρίτο, η Ευρώπη στον κόσμο και αυτό, πολύ ωραίο κεφάλαιο. Και εν συνεχεία η διαχείριση, διάρθρωση, η διοίκηση και ίσως ένα έκτο που να καλύπτει ε, το περιθώριο αποθεμάτων, ένα αποθεματικό περιθώριο ε, με, με τη στοιχείο της ευελιξίας που αναφέραμε. Ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βεβαίως και υπότιτλους Παραδείγματο χάρη στο, στο 5, στο σημείο 5 που λέει διοίκηση, να αναφέρουμε ορισμένου υποτίτλου ε, με τα στοιχεία τη ε, διαφάνειας, της, ε, 5 5α, 5β, 5γ, 5γ, δηλαδή διάφορους υπο, υποδιέρεση σε ήπια κεφάλαια υπό, τον, ε, υπό το 5. Και αυτό γίνεται. Κάτι εκεί όπου θα χρειαστούμε λιγότερη ευελιξία είναι σε ορισμένα ε, μεγάλα προγράμματα τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να περιοριστούν σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο όπως το Γαλιλαίο, στον Γαλιλαίο. Εάν δεν εξασφαλίσουμε τις πιστώσεις τις αναγκαίες θα έχουμε τη συζήτηση που γίνεται ανέκαθεν θέλουμε περισσότερες πιστώσεις, δεν υπάρχουν κλπ. Ας ε, εξασφαλίσουμε ότι ο Γκαλιλαίο θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, για το οποίο θα εξασφαλίσουμε υπό το κεφάλαιο 2, διότι περιλαμβάνει τις καινοτομίες, τους νέους κλπ, με συγκεκριμένες πιστώσεις και ότι αυτές θα είναι εγγυημένες. Να το εξασφαλίσουμε ένα εγγυημένο πλαίσιο. Όσον αφορά τώρα τη διάρκεια, όπως είπε και η Χέλγα το πρωί, δεν έχουμε ακόμα αποφασίσει, διότι τι είναι καλύτερο τα 7 χρόνια, τα 5 χρόνια. Η υπερισχύουσα άποψη υποστηρίζει την πενταετία με μία αναθεώρηση στο ενδιάμεσο ε, διάστημα. Ε, και ίσως χρειαζόμαστε μια μακροπρόθεσμη προοπτική προβλέψεων για το Ταμείο Συνοχής. Ε, γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι μάλλον η πενταετία ε, θα μας ωφελήσει περισσότερο, αλλά αυτή η συζήτηση γενικά, και έχω πέντε δευτερόλεπτα ακόμα να μιλήσω, μας έδωσε εξαιρετικά ενάψματα προς συζήτηση. Μάλιστα. Συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπες, όχι δεν θέλω μόνο τον ίσο τώρα, αλλά ε, γενικά συμφωνώ με αυτά που λες. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι το 5 5 που αναφέρει ότι θα μας δώσει πιο πολύ ευελιξία από το τα 7 χρόνια. Έχουμε εμπειρίες, δεν μας έχουν διδάξει τίποτα. Και τι μας δείχνει η εμπειρία, ότι ποτέ δεν έχουμε αυτό το review. Και αν έχουμε και συμφωνήσει με το 5 5, θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε, και εσύ ιδιαίτερα, πολύ περισσότερο από ότι εγώ, ότι θα βρεθούμε με 10 χρόνια. Δεν ε, θα αλλάξει. Το review μην περιμένετε να αποφέρει οτιδήποτε. Δεν νομίζω ότι θα είναι αντίθετη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα μας πει ότι κοιτάξτε όχι ποτέ δεν το δεχόμαστε κτλ. Ε, δεν το φαντάζομαι. Δεν ζητάει κανείς άλλος ε, το λόγο πέρα από τον Ράιμερ Μπέγκε και τον Σουζέ Μανιουέλ και την Κωνσταντζα. Και μετά δεν έχουμε κανέναν άλλον. Γάιμα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Φαίνεται στην παρούσα φάση σε ό,τι αφορά την ε, δομή του θέματος ότι θα έχει πιο πολλές τροπολογίες το θέμα αυτό από πολλές άλλες ε, εκθέσεις. Ε, φυσικά το, το πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να διακέσει τουλάχιστον πέντε χρόνια και ότι από πλευράς κατηγορία, κατηγοριών θα πρέπει να υπάρχουν ε, λίγες. Ο εισηγητής προσπάθησε να εντάξει τη στρατηγική του 2020 και των ε, υφιστάμενων ε, δομών να τα εντάξει όλα αυτά στην έκθεση. Και φυσικά αυτό μπορούμε να, μπορεί να βρει και υποστηρικτές και άλλα άτομα που δεν την υποστηρίζουν. Το θέμα είναι τι ευελιξία θα πρέπει να υπάρξει στο εσωτερικό των τομέων και μεταξύ των τομέων. Και φυσικά θα ήθελα να πω ότι το πρωτογενές δίκαιο, οι πολιτικές αναγκαιότητες που προκύπτουν από τη συνθήκη της Λισαβόνας θα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα και από εκεί ε, προκύπτουν και οι στόχοι της στρατηγικής για το 2020 και όχι αντίστροφα και μπορούμε να συζητάμε ποιες δομές ε, θέλουμε. Μου είπαν προηγουμένως ότι φυσικά και η νεολαία είναι flagship στο πλαίσιο της Ευρώπης το 2020. Μπορούμε να βάλουμε το Youth ε, in the Move. Αλλά, από την άλλη, καταλαβαίνω και αυτά που είπε ο συνάδελφος Άλβαρο ότι φυσικά και σε θέματα ελευθερίας ε, δικαιοσύνης ε, χρειαζόμαστε και μπαίνουμε σε, νέους, ε, νέες διαστάσεις και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε και πώς έχουν ενταχθεί όλα αυτά τα θέματα σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Να δούμε και η αλληλεία και το περιβάλλον και η προστασία του κλίματος μήπως θα πρέπει να μπουν σε ξεχωριστές υποκατηγορίες και σε ό,τι αφορά την αλλαγή του κλίματος και την ενεργειακή πολιτική κατά πόσο θα μπορούσαν να μπουν στο ΕΝΑΣΥ. Θα το συζητήσουμε και στο εσωτερικό της ομάδας για την δομή. Και φαντάζομαι ότι αυτό το θέμα μπορούμε να το αφήσουμε ανοιχτό μέχρι το τέλος των διαπραγματεύσεων και των συζητήσεων. Σημαντικό είναι να συζητήσουμε για τα μεγάλα project έρευνα πώς μπορεί να υπάρχει ξεχωριστή και βιώσιμη χρηματοδότηση η οποία δεν θα θέτει υπό αμφισβήτηση διαρκώς νέες προτεραιότητες. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είτε θα πούμε ναι για κάποια συγκεκριμένα μεγάλα project, τα οποία όμως θα τα χρηματοδοτήσουμε μέχρι τέλους, ή θα πούμε ότι κοιτάξτε για τον Δίνα Ιτάδε λόγο δεν μπορούμε να το χρηματοδοτήσουμε αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για θέματα ευελιξία θα πρέπει να γίνουν δύσκολε μεταρρυθμίσει στα πλαίσια τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Και αυτό που συζήτησαμε την τελευταία φορά, κάποια συγκεκριμένα ταμεία θα πρέπει να κινητοποιηθούν πάνω από το δημοσιονομικό πλαίσιο και την νομοθετική ευελιξία που ε, είναι 5% αλλά δεν το πλησιάσαμε αυτό το ποσοστό. Θα πρέπει να παραμείνουν ε, αυτές οι δυνατότητες και η ασφάλεια από το, των ειδικών ε, πολιτικών προκύπτει από, τα, από την νομική βεβαιότητα των πολιετών δημοσιονομικών προοπτικών. Η ασφάλεια πάντα είναι στην νομική βάση. Από εκεί προκύπτει. Και νομίζω ότι τα στοιχεία τα οποία ανέφερε ο Σαλβαδόρ για την ε, ευελιξία είναι συνολικά μια χαρά. Το θέμα δεν είναι μόνο να γίνεται μεταφορά από το ένα έτος στο άλλο και όχι μόνο σε έναν τομέα του προϋπολογισμού. Όχι, θα πρέπει να το συζητάμε πιο γενικά. Να υπάρχει δυνατότητα να μεταφέρονται και πιο μακροπρόθεσμα αχρησιμοποιητά κοντήλια για το χρόνο διάρκειας. Το συζητήσαμε και το ψηφίσαμε με πολύ αντιφατικό τρόπο και την προηγούμενη φορά. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να οικοδομήσουμε και κάποιες γέφυρες. Ξέρουμε ότι κάποια προγράμματα πολυετή δεν μπορούν να συνάδουν απαραίτητα με πέντε έτη. Το 5 συν 5 τώρα από τις εμπειρίες που είδαμε ε, περιορίζει υπερβολικά τον προπολογισμό και δεσμεύει το Κοινοβούλιο πέρα από την ε, τρέχουσα θητεία. Δεσμεύει του επόμενου ουσιαστικά. Γι' αυτό το να φτιάξουμε μία γέφυρα και να πούμε ότι εντάξει, επτά έτη υπό όρους και να έχουμε και τη γέφυρα, τη δυνατότητα στο μέλλον, στην επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, να περάσουμε σε πενταετές πλαίσιο και να αντιμορφωθεί με πιο δεσμευτικό τρόπο από αυτό που αναφέρεται στην έκθεση. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια λύση ενδεχομένω για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ο Σωσέ Μανουέλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια ερώτηση καταρχήν. Μιλάμε πολύ για τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Τελικά πότε ξεκινάει αυτή η στρατηγική. Γιατί στο σημείο 33 λέει ο Σιγητή ότι έχει δεκαέτη μέχρι το 2020. Εγώ δεν ξέρω αν η στρατηγική το 2020 δεν ξεκινά μόνο όταν θα υπάρχει ο υπολογισμό, Δηλαδή, μήπω ξεκινήσει την ίδια στιγμή που θα ξεκινήσουν και οι επόμενε δημοσιονομικέ προοπτικέ. Το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Πότε λοιπόν ξεκινά αυτή η στρατηγική, μήπω θα πρέπει να ξεκινήσει όταν θα υπάρχει και ο προπολογισμό, ο διαθέσιμος, κατόπιν ο εισηγητής λέει επίση ότι οι πολιτικέ που σχετίζονται με τη στρατηγική Ευρώπη 2020 θα πρέπει να ομοδοποιούνται σε ένα και μόνο τομέα, σε ένα και μόνο τίτλο. Καταλαβαίνω αυτή τη λογική, όμω, η νεολαία βρίσκεται στο τομέα 2 και όχι στην Ευρώπη 2020 ενώ ε, με σαφήνεια αποτελεί ένα στόχο της στρατηγικής, της ε, στρατηγικής Ευρώπη 2020 και όταν με σαφήνεια αποτελεί προτεραιότητα αυτής της στρατηγικής ε, αλλά και στόχο. Στο, να, θα σας πω ότι έχουμε και πέντε στόχους που αφορούν την νεολαία στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Έτσι λοιπόν Ίσως ε, θα μπορούσαμε να βάλουμε ε, α, την νεολαία στη γνώση για ανάπτυξη και την απασχόληση. Επίση, για τις δημιουργικές τομείς, μήπως ο πολιτισμός θα έπρεπε να είναι τμήμα και της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Είναι δύο αμφιβολίες που έχω εγώ. Αλλά η πεποίθησή μου είναι ότι η νεολαία πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται στην ομπρέλα της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Επίσης ε, θέλω να σας συγχαρώ που έχετε συμπεριλάβει εδώ το 4 χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση. Θεωρώ ότι κάθε δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, κάθε προϋπολογισμός θα πρέπει να βρίσκεται ε, στο πλαίσιο του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, στον προϋπολογισμό αυτό. Δηλαδή δεν πρέπει να έχουμε προϋπολογισμούς κρατικούς για εξωτερικές δράσεις, η χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση αποτελεί ένα μηχανισμό σταθερότητας χρηματοπιστωτικής και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την κοινωτική μέθοδο και να λέμε ότι όλοι οι πόροι δράσης των θεσμών θα πρέπει να εντάσσονται στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Τώρα για τη διάρκεια. Θα προτιμούσα δεκαέτη. Αν υπάρχει υποχρεωτική αναθεώρηση στα πέντε. Αυτή θα είναι η προπόθεση. Θεωρώ ότι έτσι θα είχαμε μεγαλύτερη σταθερότητα για πολιτικές όπως οι πολιτικέ συνοχής και η ΚΑΠ. Για την ΚΑΠ έχω άλλη μία αμφιβολία. Αν η κοινή γεωργική πολιτική, η κοινή αγροτική πολιτική, αντί να εντάσσεται στην αϊφόρου ανάπτυξη, μήπω θα έπρεπε και αυτή να βρίσκεται σε έναν διαφορετικό τομέα, γιατί θεωρώ ότι αποτελεί τμήμα τη ε, έξυπνη αηφόρου και καθολικής ανάπτυξης ε, και όχι μόνο στη βιώσιμη ανάπτυξη. Μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε ένα διαφορετικό τίτλο, μια αυτόνομη, έναν αυτόνομο τομέα, ένα δέλτα, δηλαδή μια γραμμή δέλτα για την κοινή αγροτική πολιτική. Επίσης, ερωτιέμαι αν μέσα σε αυτούς τους τομείς, σε αυτούς τους τίτλους, θα έχουμε και υποτομείς. Γιατί για να διατηρήσουμε λίγο λοιπόν, χάρη τη γεωργία στη βιώσιμη ανάπτυξη, αν το διατηρήσουμε αυτό, δεν ξέρουμε πώ θα πρέπει να έχουμε και έναν υποτομέα σε, στο εσωτερικό αυτού για τη γεωργία. Όπως και να έχει. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή, γιατί έχει εκπονήσει αυτή τη δομή ε, σεβόμενος τη δομή της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και το στόχους στους οποίους όλοι θέλουμε να πετύχουμε. Σας ευχαριστώ. Η Κωνσταντσε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω και να αναφέρω δύο ζητήματα. Καταρχά σε ό,τι αφορά τη δομή. Πρέπει να πω από πλευρά περιφερειακής πολιτικής ε, μας φαίνεται εξαιρετικό. Στη γνωμοδότηση ζητήσαμε η πολιτική συνοχή να περιοριστεί σε μία κατηγορία του προπολογισμού και αυτό και προτείνεται, αλλά μετά από αυτά που ακούσαμε και από τον Ράιμερ, θα πρέπει να εξασφαλίσω ότι δεν θα προσπαθήσουμε μέσα από τη δομή να πάρουμε κι, άλλες, κι άλλα ταμεία από την περιφερειακή πολιτική. Είπε, ε, Ράιμερ, να προσθέσουμε και το Ταμείο για την Αλλαγή του Κλίματος για το Περιβάλλον ναι, εγώ φαντάζομαι ότι άλλο εννοούσε, αλλά θα μπορούσα να φανταστώ ότι οι άλλοι συνάδελφοι θεωρούν ότι υπάρχει μια ευκαιρία η οποία δεν υπάρχει. Γι' αυτό λοιπόν να, να προσέξουμε τη διατύπωση προκειμένου, γιατί πιστεύω ότι τον ίδιο στόχο επιδιώκουμε, προκειμένου αυτός ο στόχος να περάσει. Σε ό,τι αφορά την διάρκεια του δημοσιονομικού πλαισίου, το είπε και ο συνάδελφος, ε, ε, υπάρχει υπάρχουν διαφορετικές ε, απόψεις και στη δική μας ομάδα. Ε, στην πολιτική την περιφερειακή θέλουμε τουλάχιστον 7 χρόνια, γιατί για μια λογική και καλή πολιτική συνοχής ε, δεν είναι λογικό να έχουμε οτιδήποτε λιγότερο γιατί με τα μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα προγράμματα δεν έχει νόημα η πενταετία. Δυστυχώς όμως πρέπει να σας δώσω δίκιο δύο φορές μία πενταετία. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι εδώ στα θεσμικά όργανα που εργαζόμαστε θα καταφέρουμε ποτέ να κάνουμε όντω ενδιάμεση αναθεώρηση. Αν ήταν αυτό δυνατόν δεν θα είχα πρόβλημα. Θα είχαμε και την συνέχεια και την σταθερότητα και την ευελιξία που θα θέλαμε με τη διάρκεια, θα το συνδυάζαμε και με τη διάρκεια της θητείας του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά επειδή δεν το πιστεύω, Εγώ πραγματικά θα αγωνιστώ για την επταετία και ευχαριστώ πάρα πολύ τον εισηγητή που το έγραψε και τόσο ξεκάθαρα μέσα στην έκθεση. Τον υποστηρίζω πλήρως και ελπίζω να καταφέρουμε να συμφωνήσουμε τουλάχιστον μέχρι το 2020 γιατί αυτό θα είχε νόημα αν η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 στο τέλος της στρατηγικής θα είχαμε και θα, μάλλον το τέλος της στρατηγικής του 2020 θα έπεφτε μαζί με το τέλος μιας επταετίας. Και δεν θα χανόμασταν για τη νέα στρατηγική την οποία θα έπρεπε ενδεχομένω να καταρτήσουμε. Άρα, με τους ε, συμμάχους πολιτικούς για την ε, περιφερειακή πολιτική θα αγωνιστούμε για την επταετία. Και πραγματικά θεωρώ την πρόταση του Σαλβαδόρ μια πολύ καλή βάση για την ε, συζήτηση. Δύο σχόλια θα ήθελα να κάνω. Καταρχάς για τη διάρκεια. Η Κωνσταντζέ μόλις είπε ότι προτιμάει τα 7 χρόνια. Αλλά αν είναι δυνατόν να υπάρξει μία ενδιάμεση έκθεση, θα μπορούσε να δεχτεί την πενταετή περίοδο. Τώρα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό λίγο περισσότερο. Τι εννοούμε με 5 χρόνια και τι εννοούμε με 5 συν 5. Συμφωνώ ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε το Συμβούλιο, να το αναθέσουμε να κάνει δηλαδή εκείνο την ενδιάμεση έκθεση ε, σε αυτήν την καθορισμένη περίοδο. Εάν όμως η βασική περίοδος του υπολογισμού είναι πέντε, αλλά ορισμένα προγράμματα είναι δεκαετή, τότε θα πρέπει να γίνει μια πραγματική ε, ε, έκθεση στο μεσοδιάστημα. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μία λύση και να εξετάσουμε αυτή την εναλλακτική. Διότι θα ήταν πάρα πολύ καλά, όπως είπε ε, και η Πρόεδρος, να συνδέεται η περίοδος του προπολογισμού με την εντολή του ε, Συμβουλίου σε ορισμένα κράτη-μέλη αυτή η διάταξη, αυτή η απόφαση θα οδηγήσει σε περισσότερα προβλήματα στον προϋπολογισμό, αλλά για μας και από απόψεως διαφάνειας είναι καλή. Όσον αφορά τώρα την ιδέα ενός άλλου τομέα ή κεφαλαίου για ε, τα αποθεματικά, εγώ πιστεύω ότι να μην έχουμε, μία, να έχουμε περισσότερη διάσπαση του προϋπολογισμού, να έχουμε υπο, υποτίτλους ή υποτομείς αν θέλετε, αλλά όχι νέους. Ε, και υπάρχει ένα υποχρεωτικό περιθώριο προϋπολογισμού. Υπάρχει ένα περιθώριο, αυτό είναι υποχρεωτικό. Ε, ποιος, για, για ποιο λόγο να έχουμε λοιπόν περαιτέρω η υποδιέρεση του περιθωρίου σε άλλους υποτομείς. Ε, ας μην περιπλέκουμε τα πράγματα περισσότερο και σκεφτούμε λίγο έξω από το κουτί. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε, εάν μπορούμε, να διαχωρίσουμε τη συζήτηση για το αποθεματικό από τη συζήτηση ε, των τομέων του προϋπολογισμού, των headings. Ευχαριστώ. Ja, möchte mich noch mal entschuldigen, ähm, dass ich jetzt gerade äh, Συγγνώμη. das Wort zu erteilen. Ε, ε, μόλις ε, συζήτησα με την Κομισιόν, κράτησε λίγο παραπάνω η συζήτησή μου, συγγνώμη, ήθελα να την φέρω μέσα στη συζήτηση, να την εμπλέξω. Λοιπόν, ε, έβαλα και τον εαυτό μου στο κατάλογο των ομιλητών, διότι βλέπω όταν μιλάμε για την διάρθρωση επανέρχονται συνεχώς δύο αντιφατικές προτάσεις, δύο αντιφατικές θέσεις. Καταρχάς η διαφάνεια, ναι εντάξει αυτή πρέπει να τη διασφαλίσουμε προς τη δημοσιότητα και τους πολίτες και αυτό είναι μία πλευρά και η άλλη πλευρά πώς μπορούμε να καταφέρουμε την ε, ύψιστη ευελιξία έτσι ώστε αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε με τον προπολογισμό να είναι εφικτό και υλοποιήσιμο. Οπότε μπορούμε να ε, φανταστούμε αυτό το οποίο ε, πρότεινε η Αν, ας πούμε το πολύ πολύ μία κατηγορία ή δύο, δύο το πολύ, εσωτερική πολιτική, εξωτερική πολιτική, που να, και όσον αφορά τις πολιτικές που ανέφερε ο Γιώραν μπορούμε να το εξετάσουμε. Εγώ πάντοτε υποστηρίζω ε, και τη διαφάνεια και την ευελιξία, παρόλο που πολλές φορές είναι σε αντίθετα στρατόπεδα. Αλλά αν έχω να επιλέξω, εγώ πιστεύω πάντοτε ότι θα διάλεγα τη διαφάνεια τη διαφάνεια. Θέλουμε να είναι διαφανείς οι ενέργειές σας. Θέλουμε οι πολίτες μας να μπορούν να ε, κοιτάξουν τον προϋπολογισμό με διαφάνεια. Αλλά τελικά το εξετάζει κανείς τον προϋπολογισμό, τον κοιτάει κανείς με το μικροσκόπιο. Ίσως ορισμένες ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις μπορεί να πάρουν ας πούμε, ένα μαγνητικό φακό και να κοιτάξουν, να εξετάσουν τον προϋπολογισμό. Ε, ποιος άλλος όμως Δεν νομίζω ότι πολλοί ασχολούνται με την εξέταση ε, του προϋπολογισμού και γι' αυτό καλό είναι να έχουμε περιορισμένο αριθμό κατηγοριών και, υποκατηγοριών. Δηλαδή, όσο το δυνατόν μικρότερος καταμερισμός. Λοιπόν, ευελιξία, θαυμάσια, πολύ ωραία ιδέα, όλα αυτά καλά και ωραία που είπαμε, αλλά αυτό που θέλω να τονίσω ξανά και που είδα ότι μελετάται από την Κομισιόν είναι πώς θα χειριστούμε τα μεγάλα έργα, τα μεγάλα προγράμματα, τα οποία πάντοτε δημιουργούν προβλήματα και σε άλλες κατηγορίες. Αυτά πιστεύω πρέπει να υπαχθούν σε μια ξεχωριστή κατηγορία. Μπορούμε να πούμε κατηγορία μεγάλων έργων, μεγάλων προγραμμάτων ε, και συναφή χρηματοδοτικά μέσα. Ορισμένοι λένε ότι χρειαζόμαστε διαφορετική μορφή χρηματοδότησης για αυτά τα μεγάλα έργα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι πρέπει όλα αυτά να τα συγκεντρώσουμε σε μια ξεχωριστή κατηγορία. Ε, ό,τι αφορά την ανάπτυξη στην κατηγορία 1, αυτό είναι σωστό, μετά μία υποκατηγορία ή ε, περαιτέρω μικρότερες υποκατηγορίες ή υποτομείς για όλα αυτά που θέλουμε να καλύψουμε στο 2020. Εμείς θέλουμε οι πολιτικές που θα υλοποιούνται στο ευρωπαϊκό επίπεδο να είναι αλληλένδετες. Και αυτό που παραδέχουμε για πρώτη φορά, ακόμα και η αγροτική πολιτική μπορεί να συμβάλλει στους δικούς μας στόχους. Δεν το πίστευα αυτό παλιά, αλλά τώρα πρέπει να το πω. Θα είναι λίγο παράδοξο, δεν λέω. Γι' αυτό πιστεύω ότι όλα αυτά αλληλοσυνδέονται υπό την κατηγορία ε, αηφόρο ανάπτυξη. Και από αυτή την κατηγορία να βγάλουμε, να αφαιρέσουμε τα μεγάλα προγράμματα. Τα πολύ μεγάλα Υπάρχουν βεβαίως και άλλα θέματα, άλλες προτάσεις που μπορούμε να μελετήσουμε. Εγώ πάντοτε είμαι υπέρ της 7 αλλά βλέπω ότι δεν με υποστηρίζουν πολύ. Δεν έχει μεγάλη πέραση αυτή η ιδέα της 7 Και εγώ τήρησα τα πέντε λεπτά, λέει η πρόεδρος. Και δεν κοίταξε και το ρολόι μου. Jetzt, ähm, hat Salvador... Ο Σαλβαντόρ έχει το λόγο. Και μετά τελειώσαμε. Η Επιτροπή τουλάχιστον. Και θα γίνει η συντάξη των συντονιστών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και αυτό που προτιμούσε ο συγητή ήταν να ακούσει πολλές ε, απόψεις και να μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτή τη συζήτηση γιατί είναι πολύ επικοδομητική. Ξεκινώντας από το θέμα της δομής της διάρθρωσης. Πράγματι, λαμβάνει η χώρα μια συζήτηση για την ευελιξία έναντι της διαφάνειας Στι ε, διάφορε κατηγορίε δαπανών. Όλα αυτά τα συζητήσαμε, ήδη τα αναφέραμε στον γράφο εργασία που παρουσιάσαμε και τη διάρθρωση. Και φυσικά, όπως είπε και η συνάδελφος Σαν ε, αν πάμε στα άκρα, χωρίς καμία κατηγορία, έχουμε τη μεγίστη ευελιξία και όσο περισσότερο φυσικά κατηγορίες και υποκατηγορίες εισαγάγουμε εδώ, τόσο Περισσότερα μέσα ευελιξίας χρειαζόμαστε σε έναν ιδανικό κόσμο. Η καλύτερη λύση ίσως θα ήταν να μην έχουμε κατηγορίες δαπανών, ε, μία διάρκεια πέντε ετών και στον τέλειο ιδανικό κόσμο δεν θα θέλαμε ούτε πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα είχαμε ετήσιο προγραμματισμό και απόλυτη ευελιξία ως κοινοβούλιο. Ξεχάστε το. Αυτό Όμω εδώ είναι κοινοτικό προπολογισμό και όχι εθνικό προπολογισμό. Και μάλιστα είναι και πολύ ενδιαφέρον αυτό ο προπολογισμό γιατί διαφέρει από οποιοδήποτε εθνικό προπολογισμό και γιατί εμεί εδώ είμαστε πολύ αξιόλογοι άνθρωποι και είμαστε και οι μόνοι που μπορούμε να κατανοήσουμε την πολυπλοκότητα του κοινοτικού προπολογισμού. Χρειαζόμαστε λοιπόν κατηγορίες δαπανών και ευελιξία. Τώρα, κοιτάξτε, εσείς ε, δικαίως ε, αναφέρατε, ορισμένοι ημών, αναφέρατε ότι θα πρέπει ο εισηγητής να είναι πιο τολμηρός, θα έπρεπε να είναι πιο τολμηρός ορισμένες από τις προτάσεις. Εγώ μπορώ να είμαι πιο τολμηρός για τις σημερινέ πολιτικές, αλλά πρέπει να παρουσιάσω μια συντηρητική δομή. Δεν μπορώ να είμαι πολύ τολμηρός, γιατί ε, αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε και αν υφιστάται αλλαγέ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Άννα Μαρία νομίζω αναφέρθηκε στα μέσα ευελιξία στο πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα περιθώρια. Ένα από τα μυστικά, ένα από τα σημεία στο οποίο μπορούμε να παρουσιάσουμε προτάσεις πολύ πιο πέρα από αυτές που ίσως είναι σε θέση να δεκτούν το, κοινοβούλιο και το, συγγνώμη, το Συμβούλιο και η Κομισιόν ε, είναι προτάσεις που έχουν να κάνουν με τη χρήση των αποθεματικών και των περιθωρίων. Εγώ ήμουν ε, κάπως πιο τολμηρός εδώ από τις άλλες τομείς, αλλά γνωρίζω ότι σε αυτή την Επιτροπή ΣΟΥΡ θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε πιο τολμηρές προτάσεις, γιατί αυτό μας ωφελεί δεν ε, σχετίζεται αυτό το θέμα άμεσα με τον όγκο των πόρων, με το μέγεθος των πόρων, ούτε με τη σύνθεση των πολιτικών, αλλά με το ότι αφορά αυτή την Επιτροπή και την Επιτροπή προπολογισμών, δηλαδή τη διαχείριση των δημοσιονομικών πόρων. Έτσι λοιπόν για το θέμα της ευελιξής νομίζω θα μπορούσαμε να πάμε πιο πέρα. Τώρα κάτι που δεν καταλαβαίνω είναι αυτή η νέα κατηγορία, η πρόταση που έγινε από κάποιον για τα μεγάλα προγράμματα. Έχουμε το Γαλιλαίο και το Ίτερ αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι το Γαλιλαίο, για το Γαλιλαίο όλοι συμφωνούν πάνω κάτω να το διατηρήσουμε και αν οι πράσινοι σκεφτούν και το Ίτερ το θεωρήσουν ως ένα μεγάλο project, ένα μεγάλο πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση των θα μπορούσαμε και να το σκεφτούμε. Τέλος πάντων είναι πολιτικό αυτό το θέμα. Δεν υπάρχουν λοιπόν τόσο μεγάλα προγράμματα για να συμπεριληφθούν σε μια υποκατηγορία. Είμαι βεβαίως ανοιχτό σε προτάσεις. Κατόπιν, μια κατηγορία για τα αποθεματικά. Είναι μια πρόταση. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε αρκετά πιο πέρα από την αρχική πρόταση του εισηγητή, αλλά το πρόβλημα να έχουμε μόνο μια κατηγορία ε, για, τα αποθεματικά, κοιτάξτε πώ θα το πώς θα το προσαρμόσουμε, ποιες είναι οι πολιτικές ε, που θα μεταφέρουν ε, ένα τμήμα των κονδυλίων που δεν έχουν δαπανηθεί εκεί. Μου φαίνεται κάπως επικίνδυνο αυτό. Ε, δεν θα ήταν και τόσο ευτυχή σε συνάδελφοι από την Επιτροπή Γεωργίας, Παραδείγματο χάρη. Αλλά είμαστε εδώ για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά το θέμα τη διάρκεια 5 ή 7 ετών. Σε έναν ιδανικό κόσμο, επαναλαμβάνω, τα 5 έτη θα μπορούσε να είναι πολύ καλά. Αλλά όσοι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, δεν είναι θέμα εμπιστοσύνη ή μη εμπιστοσύνη στο Συμβούλιο. Εντάξει, δεν έχουμε και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην ικανότητα του Συμβουλίου να κάνει μία πρόβλεψη κάθε έτη, να κάνει μία, με συγχωρείτε, μία ενδιάμεση αναθεώρηση κάθε έτη αλλά θα συμπεριλάβουμε στην έκθεσή μας ότι θα ζητήσουμε μια δεσμευτική αναθεώρηση. Εντάξει, πολύ ωραία. Ξέρουμε τι σημαίνει με αυτές τις υποχρεωτικές δεσμεύσεις που θέλουμε να επιβάλλουμε στο Συμβούλιο. Δεν είναι πραγματικά δεσμευτικές. Για το Συμβούλιο τίθεται θέμα κατόπιν ερμηνεία των συνθήκων. Αν όμως καταφέρναμε να έχουμε μία ρήτρα και ήταν διατεθειμένο το Συμβούλιο να δεσμευτεί νομικά για μια υποχρεωτική ρήτρα αναθεώρηση, τότε ναι, θα ήταν δυνατόν να σκεφτούμε άλλη διάρκεια για τι δημοσιονομικέ προοπτικέ. Όμω, βάσει τη πείρα μα αυτή τη στιγμή, γνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη γενικά χρειάζονται 7 έτη για έναν ορθό προγραμματισμό των πολιτικών του. Και εγώ νομίζω ότι προ τη στιγμή θα πρέπει να διατηρήσουμε τα 7 έτη, αν και στο μέλλον θα ήταν λογικό οι θητείε τη Κομισιόν του Κοινοβουλίου, καθώ είναι 5 έτη, να είναι αυτή η διάρκεια και των δημοσιονομικών προοπτικών. Προς το παρόν διατηρώ βέβαια εγώ τα επτά έτη. Άλλο θέμα. Τι θέλουμε να βάλουμε σε αυτή την κατηγορία της χρηματοπιστωτικής διακυβέρνησης. Θέλουμε να βάλουμε κάποιες εγγυήσεις. Έχουμε το ετήσιο πλαφόν ένα το δαπανών με την απόφαση για τους ίδιους πόρους. Ε, κοιτάξτε, θα ήθελα εγώ αυτά τα χρήματα να συμπεριληφθούν στις πολιτικές δαπανών, αλλά πρέπει να κάνουμε μια ρεαλιστική πρόταση εγώ. ήθελα αυτές οι εγγύσεις να υπάρχουν στον κοινοτικό προπολογισμό με ασφαλιστικές δικλίδες, έτσι ώστε να αποφύγουμε να χρησιμοποιηθούν αυτά τα κονδύλια για άλλες κατηγορίες δαπανών. Στην περίπτωση αυτή θα ήθελα αυτός ο μηχανισμός να συμπεριληφθεί που είναι ο μηχανισμός ε, χρηματοπιστωτική χρηματοπιστωτικής διακυβέρνησης. Θα ήθελα αυτό να τεθεί στον κοινωνικό προπολογισμό, γιατί έτσι εγγυώμαι να ε, συνεχιστεί η κοινωτική μέθοδος για την ενεργοποίησή του. Επίσης νομίζω ότι είναι ε, μια καλή συζήτηση που πρέπει να γίνει στο μέλλον μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και εντάξει θα έλεγα στους συναδέλφους ε, επί της αρχής να δεκτούμε αυτό, δηλαδή την αρχή ότι η χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη δομή των δημοσιονομικών προοπτικών. Και κατόπιν θα δούμε πώς ποσοτικοποιείται στην πραγματικότητα. Ο κ. Φερνάντες έθεσε κάποιες πολύ καλές ερωτήσεις. Πότε θα, αρχίσουμε, πότε θα αρχίσει να τρέχει η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 για μας ξεκινά το 2014. Έτσι λοιπόν αυτή η δομή της στρατηγικής κατά την απόψή μου ξεκινά το 2014 και τώρα για την νεολαία. Τα τμήματα που αναφέρονται στην απασχόληση και φυσικά έχουν να κάνουν με την νεολαία θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην κατηγορία στρατηγική Ευρώπη 2020. Και εγώ στην κατηγορία της ηθαγένειας είχα βάλει τα θέματα της νεολαίας και του πολιτισμού γιατί θεωρώ ότι έχουν να κάνουν με την συμμετοχή των νέων την ένταξη των νέων στα συμμετοχικά μοντέλα στην κοινωνία. Έτσι λοιπόν εδώ θα προτιμούσα να τα αφήσω τους νέους στην ηθαγένεια μαζί με τον πολιτισμό. Τώρα, ας επιστρέψουμε στην ιδέα με της ε, σταθερής φωτογραφίας. Ωστόσο ζητούσαμε, συνειδητοποίησα ότι στο γενικό τομέα της πρώτης κατηγορίας θα πρέπει να έχουμε απλώς Ευρώπη 2020. Και επίσης σκέφτηκα ότι ο πολιτιστικός ε, τομέας, πολιτιστική βιομηχανία, τα οπτικοκουστικά συγκεκριμένα, πιθανότατα θα έπρεπε να είναι στην γνώση για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Βλέπετε μία τόσο ανοιχτή συζήτηση, βοήθεια για να σκεφτούμε κάποιες αλλαγές στην αρχική φωτογραφία. Δηλαδή ο εισηγητής ε, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να σας πει ποια θα είναι η οριστική δομή. Όσο περισσότερο συζητάμε, τόσο περισσότερες οπτικές ε, έρχονται στο νου μου και όλα μου φαίνονται αποδεκτά. Στο τρίγωνο της γνώσης, ε, έρευνα, καινοτομία και εκπαίδευση, θα ε, ήθελα να μπει σε αυτό το ένα α σε αυτή την υποκατηγορία. Νομίζω ότι εκεί έγκυται ο πυρήνα τη ανταγωνιστικότητα τη Ευρώπη για το μέλλον. Όλε οι υπόλοιπε πολιτικέ που συνοδεύουν αυτή την κατηγορία 1α τελικά έχουν πολύ μικρή ποσοτικοποίηση στον προπολογισμό, αλλά εγώ νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στην κατηγορία 1α. Όπω και να έχει, είμαι ανοιχτό οποιαδήποτε πρόταση Στην έκθεση υπάρχουν λίγες θέσεις κατηγορηματικές. Βεβαίως και είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση και στην ανάλυση νέων προτάσεων. Και για τη δομή αυτή, όπως και για την ευελιξία. Αλλά πιστεύω ότι το έγγραφο εργασία χρησιμεύσε για να ξεκινήσει η συζήτηση στι διάφορε πολιτικέ ομάδε και αυτό ακριβώ θέλουμε να πετύχουμε. Είμαστε ακόμα στην αρχή μια περίοδου κατάθεση τροπολογιών και στη συνέχεια θα υπάρξουν ε, προφανώ και συμβιβαστικέ τροπολογίε. Έχουμε ακόμη πολύ χρόνο για να εμπλουτίσουμε τη δομή και να την προσαρμόσουμε στις ανάγκες για να πετύχουμε και τι 500 ψήφου. Ja, in der Tat, das haben wir. Ναι, όντω ε, έχουμε χρόνο. Τώρα, αν ε, στα διάφορα δεν υπάρχει κάτι άλλο, Να σας ανακοινώσω μόνο ότι η επόμενη συνεδρίασή μας θα λάβει η χώρα στις 17 Απριλίου. Συγγνώμη, στις 7 Απριλίου, στο Στρασβούργο. Και τώρα να παρακαλέσω τους συντονιστές να μένουν στην αίθουσα. und die anderen Saal zu verlassen. Και οι υπόλοιποι παρακαλώ να φύγουν.